ε, για αυτού του εργαζομένου Βουλγαρία και Ρουμανία και αυτή η ημερομηνία ήταν, είναι η 31η Δεκεμβρίου του 2011. Οπότε παρακαλώ λάβετε υπόψη αυτό, συνάδελφε, και στηρίξτε αυτό το βήμα. Ναι, ναι, ναι, λέει ο πρόεδρο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα μία παρατήρηση, μάλλον μία παρέμβαση υπέρ τη πρόταση. Είναι υπέρ. Ναι, ναι, ναι, ναι, υπέρ. Ευχαριστώ, πρόεδρε.